είναι σαν να παραβαίνει την εθνική κυριαρχία και των υπολείπων 26 χωρών που έχουν συμφωνήσει για αυτή τη συνθήκη. Και να πω και ένα ακόμα πράγμα. Η πλειοψηφία των δύο τρίτων ε, προέκυψε από μια πλειοψηφία 50% μόνο σε ψήφους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση συντάγματος θα πρέπει να εξασφαλίζει ευρεία συνένεση στο λαό. Αυτή τη στιγμή όμω, δεδομένου ότι είναι μόνο μια πολιτική δύναμη που έχει αυτή την πλειοψηφία, δεν εξασφαλίζει αυτή την συνένεση. Δηλαδή, κατά βάση, σεβόμαστε το γράμμα, αλλά παραβαίνουμε το πνεύμα τη συνένεση. Ευχαριστώ. Κύριε Ταβάρη, διαδικασία μπλε κάρτα τη δέχεστε? Okay, so please. Λοιπόν, ερώτηση. Ποιος σας έχει δώσει το δικαίωμα να μιλάτε έξω ονόματος των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Έγινε μια έρευνα η οποία απέδειξε ότι πολλοί από αυτούς τους πολίτες δεν